Συνεχίζουμε λοιπόν. Με ενημέρωσαν κυρίες και κύριοι ότι κατά τον ε, τρίτο γύρο προέκυψε ένα επεισόδιο στις ε, κάλπες. Ένας ευρωβουλευτής αρνήθηκε να δείξει τη ταυτότητά του. Οι ψηφολέκτες λοιπόν ε, διαμαρτυρήθηκαν, συζήτησαν, συναντήθηκαν, συζήτησαν μεταξύ τους και αποφάσισαν την ψήφο αυτή και το ψηφοδέλτιο αυτό να το κρίνουν άκυρο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν σας ζητήσουν οι ψηφολέκτες να δείχνετε την ταυτότητά σας ή το διαβατήριό σας, να το πράτετε. Έρχομαι λοιπόν στο αποτέλεσμα της, ε, του τρίτου γύρου ψηφοφορίας. 719 ψήφισαν, 29 άκυρα, έγκυρα ψηφοδέλτια, 690. Η απόλυτη πλειοψηφία ως εκ τούτου είναι 346 ψήφοι. Κυρία Φορέντσα, 45. Λαμπέρτ, 53. Πιτέλα, 199. Ρεμπέγκα, 44 ψήφους. Στίβενς, 58. Ο κύριος Ταγιάννη. 291 ψήφοι. Επειδή λοιπόν κανένας υποψήφιος δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία, ε, θα περάσουμε στον τέταρτο γύρο ψηφοφορίας και με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού Κατά τον τέταρτο γύρο θέτουν υποψηφιότητα μόνο οι δύο εκείνοι υποψήφοι οι οποίοι κατά, την, κατά τον τρίτο γύρο ψηφοφορίας έλαβαν το μεγαλύτερο σύνολο ψήφων. Και προηγούνται λοιπόν ο κύριος Πιτέλα και ο κύριος Ταγιάννη. Τα ονόματα τα ανέφερα με αλφαβητική σειρά. Διακόπτεται λοιπόν τώρα η συνεδρίαση μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ και θα επανέλθουμε στις 9.21. Ευχαριστώ πολύ.